Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Παρακαλώ καθίστε Ησυχώ Έλαβα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες αιτήματα διορισμού στις επιτροπές και αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος θα εγγραφεί στα πρακτικά της Συνόδους και εάν ε, δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Η ΙΜΚΟ και ΕΚΟΝ διαβίβασαν τρεις, τρία διορθωτικά κείμενα. Τα δύο της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, συνοδεύονται από μία δήλωση και υπάρχουν στην ιστοσελίδα τη Συνόδου On Direct και συνεπώς οι δηλώσεις θα εγγραφούν στα πρακτικά. Δυνάμει του άρθρου 216 αυτά τα ε, σημειώματα και οι δηλώσεις θα εγκριθούν εκτός και αν στις 24 ώρες μια πολιτική ομάδα ή 40 ε, ε, μέλη ζητήσουν να γίνει ε, να εγκριθεί κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και μία πρόταση του κυρίου Λάμσντορφ για την 68η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση αυτή θεωρείται ότι εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες και αρχίζουμε με την απλοποιημένη διαδικασία, άρθρο 138, έκθεση Ντότς για τα αποθέματα γάδου. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, ποιοι μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία για την έκθεση Dodge. Le vote est clos. Πέρας. Κλείνει τώρα. Όχι, όχι, μπορείτε να ψηφίσετε, μπορείτε να ψηφίσετε. Εγκρίνεται η έκθεση. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση με την ίδια δικασία, την έκθεση Wickstrom για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Γιάσεκ Όλκιτ Κούρσκι. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχέσε εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση με την ίδια διαδικασία του κ. Στογιάνοφ για την αίτηση άρσης της ασυλίας της Μαλγκοζάτα Χάνσλικ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Λίχτενμπέργκερ για την αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας του Αλεξάνδερ Άλβαρο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις εκθέσεις Γκαρσές Ραμών για το νέο θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Καταναλωτών. Ψηφίζουμε με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Le vote Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Τσφίχκα για το ευεργέτημα παινία σε δια... συνοριακές διαφορές επιαστικών και εμπορικών υποθέσεων. Ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, σε δεύτερη ανάγνωση, θα δούμε την τελωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία, άρα Θεωρούμε ότι εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Στη συνέχεια και σε δεύτερη ανάγνωση θα δούμε τη θέση ε, του Συμβουλίου σε σχέση με τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικού ιατρικούς σκοπούς. Η τροπολογία 6 έχει αποσυρθεί. Πρόκειται για την έκθεση ΡΙΣΕ, τροπολογία 1, με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Με ονομαστική αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται και τέλος ε, τροπολογία 2. Με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Καμία τροπολογία δεν εγκρίθηκε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η θέση του Συμβουλίου εγκρίνεται. Να συγχαρούμε την κυρία Ρης. Στη συνέχεια ψηφίζουμε την έκθεση Μωρένα Σαρτιέ για τις αλέχιστες απαιτήσει υγείας και ασφάλειας αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προηγούμενους από φυσικούς παράγοντες. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια ψηφίζουμε το σχέδιο DOTS ε, για τα αποθέματα γάδου και αλλιευτικές δραστηριότητες. Εξετάζουμε την πρόταση κανονισμού και αρχίζουμε με ένα μπλοκ τροπολογιών 19 της Επιτροπής Αλίας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεν είναι σαφές, γι' αυτό θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία για τις 19 τροπολογίες της Επιτροπής Αλίας. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν. με μεγάλη, εγκρίνονται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Θέλετε να επαληθεύσουμε, εντάξει, ελέγχουμε για την 7, αρχίζει η ψηφοφορία, ηλεκτρονική για την τροπολογία υπαριθμών 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να επαληθεύσουμε βεβαίως. Τροπολογία 17 αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ωραία. Θαυμάσια. Πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με, ε, με ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στην έκθεση για Κολίνο, για την, το έγκλημα διαφθορά κλπ. Εγκληματικές δραστηριότητες. Παράγραφος 3 επί του αρχικού κειμένου, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Αν θέλετε να επαληθεύσουμε για την 7, αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν είναι όμως απόλυτα σαφές. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία υπαριθμών 8 ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 19 και ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 21 ε, τροπολογία 4 υπέρ Υπέρ, υπέρ της 4. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρ το αρχικό κείμενο με τρεις ξεχωριστές ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και με ονομαστική το δεύτερο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική αρχίζει η ψηφοφορία. πέρας και απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο αρχικό κείμενο, παράγραφος 43, με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Πέρας Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 53, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 55. Το αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 58. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 80. Δύο τμήματα. Πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 81, αρχικό, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 93, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 96. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να το ελέγχουμε αν και μου φαινόταν ξεκάθαρο.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 Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε λοιπόν. Τροπολογία 6. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην παράγραφο 106, αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 107, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 108. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 124. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 127. Ελέγχουμε. Εντάξει. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 127 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 128 επίσης ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, μετά την παράγραφο 128, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 129 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 130. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 133 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 139 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται παράγραφος 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 141 με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 144, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα η αναθεωρημένη τροπολογία 3, ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Την 3. Αναφερμένη 3. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Στο recital πύλα την εικόνα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται BH λατινικό, πρώτο τμήμα ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. BK Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εκλού. Ε, le B. Απορρίπτεται. BL σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. B, π, λατινικό, με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα της πρώτης ψηφίσματος, ψήφι περ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε το λόγο κύριε Σιγητά. Κύριε να έχετε το λόγο. Πού είστε όμως, σας βλέπω. Μάλιστα, σας είδα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Γιακολίνο. Ah, ça ne marche pas. Αν πατώντας το κουμπί δεν ανάβει το μικρόφωνο, περάστε στο διπλανό. Ah, oh, voilà. ringraziare tutti... επιτέλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στην ε, Επιτροπή ε, που ε, ε, μας επέτρεψαν να φτάσουμε στο στάδιο αυτό στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανομών εξόδων. Έτσι έχουμε εντολή να υποβάλουμε κατευθυντήριες γραμμές στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να αναλάβουν τον αγώνα κατά αυτής της μορφής εγκλήματος. Προφανώς είναι πολύ σημαντική αυτή η ευρωπαϊκή εντολή καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Διακόπτουμε μέχρι τις 12.30 τώρα. Θα τα πούμε αργότερα για τις ψηφοφορίες.